E, Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι η συνεδρίαση συγκροτήσεως σε σώμα της Επιτροπής για τη νέα θητεία 2009-2013. Άλλο 2014. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή μας υπάρχει μόλις για δεύτερη θητεία. Κατά το παρελθόν η Επιτροπή μας αποτελούσε ένα τμήμα της Επιτροπής Μεταφορών. Οπότε έχουμε πέντε χρόνια εμπειρίας σαν εντελώς ανεξάρτητη Κοινοβουλευτική Επιτροπή και σήμερα ξεκινάμε άλλη μια θητεία του κοινοβουλευτικού αυτού οργάνου. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που προεδρεύω αυτού του τμήματος της ε, συνεδριάσεως και αυτό διότι ο πρόεδρος και, πρώτη, και ο πρώτος αντιπρόεδρος απουσιάζουν. Εγώ ήμουν δεύτερος αντιπρόεδρος και έτσι έχω την τιμή σήμερα να προεδρεύσω του πρώτου τμήματος της συνεδριάσεώς μας. Θα μιλήσω τώρα αγγλικά, θα ήθελα σε ενημερώσω για κάποια πράγματα. Να υπενθυμίσω ποιο είναι ο σκοπό τη συνεδριάσεω. Η συγκρότηση σε σώμα του Προεδρείου. Και επίση θα γίνουν οι εκλογέ. Πρώτα πρέπει να κλέξουμε τον Πρόεδρο και μετά τους Αντιπροέδρους. Να σας υπενθυμίσω ότι σύντομα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό αν υπάρχει ένας υποψήφιος για μία θέση, βεβαίως υπάρχει πιθανότητα εκλογής διαβοής. Υπάρχει και άλλη πιθανότητα. Αν κάποιος επιθυμεί μυστική ψηφοφορία, θα πρέπει να ζητήσουν οκτώ βουλευτές την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Αυτό ισχύει και για τον Πρόεδρο και για τους Αντιπροέδρους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις εκλογές μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την απαρτία. Θέλουμε να δούμε αν είναι νόμιμη ψηφοφορία για ένα νέο πρόεδρο της Επιτροπής. Αν έχουμε απαρτία η γραμματεία μπορεί να μου επιβεβαιώσει ότι έχουμε απαρτία. Μου λένε λοιπόν ότι έχουμε απαρτία. Μπορούν να διεξαχθούν οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο. Τώρα, στην επόμενη φάση της διαδικασίας θα ζητήσουμε υποβολή υποψηφιωτήτων για τη θέση του Προέδρου. Ποιο μέλος πολιτικής ομάδας θα προτείνει υποψήφιο για τη θέση Προέδρου, ο κύριος Φανλίστερ Ρόε, όπου είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σας ευχαριστώ Προέδρε, με τα χαράς να το κάνω αυτό. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική και όπως είπατε ε, μπαίνουμε στη δεύτερη θητεία μας και εκ μέρους του ΕΛΚ έχω να προτείνω την κυρία Χούμπνερ είναι νοεκλεγήσα στο Κοινοβούλιο, αλλά έχει εξαιρετικά προσόντα. Κυρίως στον τομέα με τον οποίο ασχολούμαστε και πιστεύω ότι μπορεί να προωθήσει τις εργασίες μας και να μας βοηθήσει. Η ομάδα λοιπόν του ΕΛΚ θέλει να προτείνει την κυρία Ντανούτα Χούμπνερ να είναι πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό θα πρέπει να ζητήσω από τον υποψήφιο ή την υποψήφια σε αυτή την περίπτωση να επιβεβαίωσει την υποψηφιότητά της. Ναι, λέει η κυρία Χούμπνερ, συμφωνώ. Είμαι υποψήφια. Ευχαριστώ. Συμφωνεί λοιπόν η υποψήφια. Κάναμε ό,τι επιθυμεί ο εσωτερικό κανονισμό. ό,τι προβλέπει. Υπάρχουν παρατηρήσεις, υπάρχουν άλλε προτάσει, άλλε υποψηφιότητε για τη θέση του Προέδρου. Πολιτικός είναι δυνατόν. Θα πρέπει βέβαια να μιλήσει κάποιο μέλος πολιτικής ομάδας. Σχόλια, ορίστε, παρακαλώ να μας πείτε ποιος είστε. Φρανσουά Αλφονσί, για τους πράσινους. Συμφωνούμε με αυτά που πρότεινε η ομάδα, με την υποψηφιότητα του ΕΛΚ, συμφωνούμε στα πλαίσια Γενική Συμφωνία. Ένα ερώτημα. Η κυρία Χούμπνερ ήταν Ευρωπαία Επίτροπος μέχρι τώρα. Το πρώτο, τα πρώτα χαρτοφυλάκια τα οποία θα πρέπει, με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αυτά με τα οποία ασχολείται όταν ήταν Επίτροπος. Μήπως υπάρχει πρόβλημα επικάλυψης καθηκόντων όσον αφορά αυτά τα χαρτοφυλάκια που, που, που είχε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Να θέσω το ερώτημα στην κυρία Επίτροπο να απαντήσει σε αυτό το σχόλιο, σε αυτή την παρατήρηση. Αν έχει την καλοσύνη, απαντήστε μας. Δεν είμαι ακόμα πρόεδρος της Επιτροπής, άρα δεν μπορώ να κάνω πρόταση για το συγκεκριμένο θέμα που ετέθη, αλλά φαντάζομαι ότι, εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε τέτοια σύγκρουση, ενδεχόμενο συγκρούσεως συμφερόντων, μπορεί να εξευρεθεί η λύση. Και στην περίπτωση της ακροάσεως αν εκλεγώ και αν είμαι πρόεδρος της Επίτροπης θα μπορούσα να ζητήσω από κάποιους από τους ε, αναπληρωτές μου να με αντικαταστήσει. για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των συναδέλφων των Πρασίνων. Πιστεύω ότι όταν γίνεται κανείς μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όταν προεδρεύει αυτής της Επιτροπής, αυτό καθε αυτό δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει τέτοια υπόνοια ή αν υπάρξει τέτοια υπόνοια, πιστεύω ένθερμα ότι αν κάποιος σέβεται τους κανόνες, δεν μπορεί να προκύψει τέτοια κατάσταση. Πιστεύω ότι θα βρούμε και λύσεις στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο ανέφερε ο συνάδελφός μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Άλλα σχόλια ή παρατηρήσεις παρακαλώ. Ωραία, δεν υπάρχει πρόταση για μυστική ψηφοφορία, οπότε εκλέγεται η υποψήφια ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Uh, Καλώς. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή τη συνεδρίαση και το επόμενο καθήκον μας είναι να οργανώσουμε την εκλογή των τεσσάρων αντιπροέδρων μας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει αλλάξει η απαρτία στο μεταξύ, οπότε δεν χρειάζεται να ελέγξουμε και πάλι την απαρτία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ε, ζητώντας από εσάς να μου πείτε κατά πόσο έχουμε κάποιον υποψήφιο για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής αυτής. Παρακαλώ. Η κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χούπνερ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ελπίζω ότι θα είσαστε μια καλή πρόεδρος και ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Ελπίζω επίσης ότι το πέρασμά σας από την Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην είναι τόσο δύσκολο και ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πάνω στις μελλοντικές διαρθρωτικές πολιτικές για την Ευρώπη. Εγώ προτείνω τον κύριο Γιώργο Τραβακάκη ως πρώτο αντιπρόεδρο και Πιστεύω ότι θα είναι ένας πρώτος αντιπρόεδρος εξαίρετος. Έρχεται από την Κρήτη. Έχει ασχοληθεί πολύ με τα θέματα τα διαρθρωτικά και αυτή είναι η πρότασή μας για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Κύριο Σταυρακάκης, λοιπόν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταυρακάκης, λοιπόν, λέτε ότι προτείνεται, αν συμφωνεί, Παρακαλώ κύριε Σταυρακάκη. Ναι, αποδέχομαι την υποψηφιότητα και ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Η επόμενη όμως ερώτησή μου είναι υπάρχει άλλος υποψήφιος για τη θέση αυτή του πρώτου αντιπρόεδρου. Όχι από ό,τι βλέπω. Συνεπώς μπορούμε, φαντάζομαι, να ψηφίσουμε διαβοήση. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να πω ότι από όλους τους υποψηφίους έχουμε πάρει τη δήλωση οικονομικών τους συμφερόντων. Πρέπει να το ξέρετε δηλαδή ότι όλες οι προϋποθέσεις καλύπτονται για τις εκλογές αυτές. Συνεχίζουμε λοιπόν και τώρα Παρακαλώ να μου πείτε αν υπάρχει υποψήφιος για τη θέση του δευτέρου αντιπρόεδρου, παρακαλώ, της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, ο κύριος Βανιστερόη. Πρόεδρε, χαίρομαι που αναλάβατε την Προεδρία. Αμέσως θα σας πω τον υποψήφιό μας για τη θέση του δευτέρου αντιπρόεδρου. είναι ο Μάρκος Πίπερ. Αυτόν προτείνουμε. Ευρωβουλευτής έχει ασχοληθεί με τα θέματα της Επιτροπής αυτής και στην προηγούμενη θητεία. Ο Μάρκος Πίπερ λοιπόν είναι ο υποψηφιός μας για την δεύτερη αντιπροεδρία παρακαλώ. Πρόεδρος, ωραία. Ο Μάρκος Πίπερ να μας πει κατά πόσο συμφωνεί να είναι υποψήφιος για τη θέση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ σας συγχαίρω πρώτα απ' όλα για την εκλογή σας και δέχομαι ευχαρίστω την υποψηφιότητα αυτή. Καλώς, ωραία. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα για τη θέση του Δευτέρου Αντιπροέδρου, παρακαλώ. Όχι από ό,τι βλέπω, οπότε πάλι εψηφίζουμε διαβοής. Παρακαλώ τον κύριο Μάρκο Πίπερ να έρθει εδώ στο Προεδρείο, να καθίσει δίπλα μα. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο σημείο που είναι η εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Και εδώ πάλι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στα χαρητήρια για τη νέα σας θέση στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να πω ότι η ομάδα του Άλτα υποστηρίζει την κυρία Χουσμάνοβα για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Η κυρία Χουσμάνοβα ήταν μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης την προηγούμενη θητεία. Ήταν και τότε αντιπρόεδρος και η ομάδα μας την υποστηρίζει δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα λόγω προσωπικού προβλήματος, ζητά συγγνώμη γι' αυτό και μου ζήτησε να σας πω ότι δέχεται την υποψηφιότητα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δήλωση. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για την θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Εάν δεν υπάρχουν, ξανά διαβοής μπορούμε να επικυρώσουμε και αυτή την εκλογή. Και πάμε στην τελευταία ψηφοφορία για τη θέση του τέταρτου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει υποψήφιος για αυτή τη θέση. Ορίστε. Ναι, κυρία Πρόεδρε, η ομάδα των Βασίνων προτείνει τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο, που είναι Έλληνας, που από τη Θεσσαλονίκη και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα προβλήματα των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Δράτω με της προτάσεως αυτής της στιγμής που παίρνω το λόγο να συγχαρώ κυρία Πρόεδρε και εύχομαι μια υπέροχη θητεία σε εσά και στο Προεδρείο σας. Thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσουμε τον κύριο Τρεμόπουλο αν συμφωνείτε να είστε υποψήφιος για αυτή τη θέση. Με τη σειρά μου σας συγχαίρω που εκλεγήκατε στη θέση της Προέδρου και του συναδέλφους αντιπροέδρους και αποδέχομαι την πρόταση. It takes some time to get it. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για τη μετάφραση των ελληνικών. Ευχαριστώ για τη δήλωσή σας, λέει Πρόεδρος. Υπάρχει άλλος υποψήφιος για αυτή τη θέση. Αν δεν υπάρχει, μπορούμε ξανά διαβοή, να επικυρώσουμε και αυτή την εκλογή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για αυτή την γρήγορη διεκπαιρέωση της διαδικασίας και θα ήθελα δύο λεπτά από το χρόνο σας για να σας ευχαριστήσω. Το εκτιμώ. Εκτιμώ πάρα πολύ την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Ε, θα είμαι προσβάσιμη, θα είμαι αποτελεσματική, θα είμαι παραγωγική πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Σίγουρα θα πρέπει να συνεργαστούμε για να πετυχαίνουμε συνένεση έναντι των κοινών προκλήσεων και των κοινών οραμάτων μας. Θα πρέπει να συνεργαστούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Θα οικοδομήσουμε πάνω στα επιτεύγματα αυτής της Επιτροπής, στα επιτεύγματα του παρελθόντος. Εργάστηκε σκληρά αυτή η Επιτροπή κατά τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε μόνο πολιτική συζήτηση που θα είναι κρίσιμη σημασία στα επόμενα χρόνια, αλλά επίσης θα γίνει και συγκεκριμένη δουλειά. Θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα από αυτή την Επιτροπή. Και δεσμεύομαι να υπερασπιστώ τις θέσεις μας, όσα υποστηρίζουμε. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να δημιουργήσω δημιουργικό πνεύμα για την Επιτροπή μας. Για μία ακόμη φορά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην ε, τακτική μας συνεδρίαση, στην κανονική μας συνεδρίαση, οπότε επισήμως λύγει αυτό το τμήμα της συνεδριάσεως. Η συνεδρίαση συγκροτήσω σε σώμα έληξε και τώρα ξεκινάμε στην τακτική μας, τακτική μας συνεδρίαση και έχουμε ένα σχέδιο ημερήσιας διάταξης το οποίο διανεμήθη και το σχέδιο μερίσιας διάταξης το έχετε στη διάθεσή σας. Το πρώτο σημείο βέβαια είναι η έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης για αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν λάβαμε κάποιες προτάσεις τροποποίησεως του σχεδίου ημερησίας διατάξεως. Αν λοιπόν δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα τώρα, εγκρίνεται ως έχει, ως διενεμήθη η ημερησία διάταξη. Θέλετε κάποια αλλαγή? Όχι. Δεν χρειάζεται αλλαγή μερίσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Ας σας πω ότι και τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Επιτροπής της 16ης Απριλίου διανεμήθησαν μόλις τώρα προς ενημέρωσή σας. Διότι σαν νέο κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να τα εγκρίνουμε. Έχουν διανεμηθεί προς ενημέρωσή σας τα πρακτικά και μπορούμε να πάμε στο σημείο παριθμών 3 της ανακοινώσης του Προέδρου. Ανακοινώσει της Προέδρου μάλλον, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα. Έχω τρία θέματα στις ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι σχετικά με την γνωμοδότηση του προπολογισμού, που είναι κατεπήγον θέμα για τις επόμενες εβδομάδες να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε διορίσει συντάκτη για την γνωμοδότηση για τον προπολογισμό του 2010. Την κυρία Πέτσα από το ΕΛΚ δεν επανεξελέγει όμως, οπότε έχουμε αυτή την πρόκληση. Λέω πρόκληση διότι το χρονοδιάγραμμα είναι άκρος περιορισμένο. Πρέπει να εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό, αλλά χρειαζόμαστε συντάκτη για τη γνωμοδότηση. Και ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ περιορισμένου χρονικού ορίου όταν τα θέματα δεν είναι επίμαχα, η πρόεδρος κανονικά προτείνεται ως συντάκτης, συντάκτρια του κειμένου. Και αυτή την πρόταση σας κάνω τώρα. Συμφωνείτε η πρόεδρος της Επιτροπής να είναι συντάκτρια για την γνωμοδότηση για τον προπολογισμό του 2010. Αυτό είναι το ερώτημα που σας απευθύνω. Ναι, Λαμπέρ. Ευχαριστώ κυρία. Ευχαριστώ πράγματι. Σωστά τα είπατε. Ε, δεν πρόκειται περί εκλογής ε, εδώ πέρα, αλλά πράγματι εμείς ε, δίνουμε απλά την ε, άποψή μας όσον αφορά τον προϋπολογισμό, την οποία μετά παίρνει η πρόεδρος υπομάλης και εξηγεί ότι πρόκειται για την ε, άποψή μας. Διαβάζοντας λοιπόν εδώ πέρα το σχετικό έγγραφο ε, βλέπω ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι υπογραμμισμένο. Υπάρχουν κάποια Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία είναι προς ε, ανανέωση. Λαμπέρ, να σε διακόψω γιατί θα το συζητήσουμε αυτό ούτω ή άλλω. Είναι το σημείο 5 στη μερίσια διάταξη. Το θέμα τώρα είναι αν συμφωνούμε στον εισηγητή. Ναι, ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Θα πω αυτό που είχα να πω αργότερο. Σα ευχαριστώ. Τίποτα άλλο επί τη διαδικασία. Ναι, παρακαλώ, κυρία Σωτό. Ähm, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, κάνατε μία δήλωση ήδη, είπατε πως εκεί όπου υπάρχουν συγκροώμενα συμφέροντα πρέπει αυτό να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. Βεβαίως εδώ πέρα ο προπολογισμός είναι ένας προπολογισμός που από την ε, Κομισιόν και εσείς ε, το θεωρούν προβληματικό να τον ε, δεχτούμε έτσι και να Ναι, το χειριστείτε εσείς. Νομίζω καλύτερα θα είναι να πάει σε έναν αντιπρόεδρο ή στην ε, κοινοβουλευτική ομάδα. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αν θέλετε να προτείνετε τον πρώτο αντιπρόεδρο, ευχαρίστω. Κάποιο άλλο σχόλιο από αυτό. Um, ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την δική μας ομάδα πράγματι εμείς υποστηρίζουμε την πρόεδρο να το αναλάβει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα γιατί τουλάχιστον πέρσι και πρόπερσι στη συζήτηση του προπολογισμού δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα μεταξύ ημών και της ε, Κομισιόν. Από κοινού εμείς και η Κομισιόν είχαμε πρόβλημα με το Συμβούλιο. Οπότε δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποιο πρόβλημα συγκρόμενων ε, συμφερόντων. Θα ήθελα να πω δε στον κύριο Στελερό ότι τα πιλωτικά έργα που είχαμε τα τελευταία χρόνια πρέπει να επανεισαχθούν εδώ πέρα να υπάρχει εγγύηση γι' αυτό και για τον φετινό προπολογισμό του 2010 δηλαδή, γιατί είναι διετή τα πιλωτικά έργα και πρέπει να προβληθούν βέβαια οι απαραίτητε δαπάνε. Πράγματι θα γίνει συζήτηση στο σημείο 5 όπως σας είπα Τώρα όμω έχουμε την ε, πρόταση τη κυρία Δεν ξέρω αν ε, κάποιο άλλο θέλει να σχολιάσει αυτή την πρόταση. Please. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι ο εισηγητή για τον προπολογισμό του επομένου έτου και υπ' αυτή την ιδιότητα ως ένα ταπεινό αναπληρωματικό μέλος τη Επιτροπή. θα ήθελα να υπογραμμίσω πώ η συζήτησή μας και το πρόβλημά μας είναι με το Συμβούλιο. Ε, εκεί εμείς τροποποιούμε το σχέδιο προϋπολογισμού και το προσχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό υλικό ως υπόβαθρο, οπότε δεν βλέπω εγώ κάποιο πρόβλημα ότι ε, να αναλάβει αυτό το έργο η πρόεδρος τη Επιτροπής μας και ο αρμόδιος Επιτροπός. Πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί του προσχεδίου αυτού του υπερπολογισμού και Επισήμω βεβαίω, αντικείμενο τη συζήτησή μα είναι το σχέδιο προπολογισμού που υπέβαλε αρχέ Ιουλίου το Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο. Άλλα σχόλια. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα την κυρία Στέτερα αν επιμένει στην άποψή της. Ναι, εντάξει, τότε θα το συζητήσουν οι συντονιστές. Αμέσως μετά θα το συζητήσουμε το θέμα. Παρακαλώ. Ναι, εμείς ως πράσινοι επιμένουμε στη θέση μας. Μάλιστα, οπότε πάει στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών αυτό το θέμα που θα ακολουθήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα τώρα να συγνωστοποιήσω πως ε, η προθεσμία για τροπολογίες ξεκινάει από σήμερα και είναι μέχρι τις 10 Αυγούστου. Η ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης θα γίνει στην συνεδρίασή μας στις 2 Σεπτεμβρίου γιατί πιέζει ο χρόνος. Οπότε συμφωνήσαμε να δούμε το ζήτημα του ή της εισηγητού και της Προέδρου στην ε, συνεδρία των συντονιστών. Η δεύτερη ανακοίνωσή μου στο σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης αφορά την ακρόαση του νέου Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής. Ίσως γνωρίζετε πως η διάσκεψη των Προέδρων σε 9 Ιουλίου συμφώνησε σε μια πιο ευκίνητη διαδικασία για αυτές τις ακροάσεις και ο προτινόμενος επίτροπος θα εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής μας στις 2 Σεπτεμβρίου και κατόπιν θα ακολουθήσει μια συνεδρίαση των συντονιστών οι οποίοι θα αξιολογήσουν την ακρόαση και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συντονιστών θα παρουσιαστεί στην διάσκεψη των πρόεδρων του Κοινοβουλίου και μάλλον εκεί θα τελειώσει ο δικός μας ρόλος. Η υπερψήφιση ή μη της Επιτροπής θα γίνει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο για το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω αφορά τα έγγραφα που έχετε μπροστά σας. Έχετε ένα εγχειρίδιο για την πολιτική συνοχής και την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και πολλές σημειώσεις που θα βρείτε ε, θα βρείτε χρήσιμες ελπίζω. Είναι στα αγγλικά αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας μοιραστούν και μεταφράσεις ε, ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Θα βρείτε λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ε, νέους και τις νέες βουλευτές στην Επιτροπή μας, θα βρείτε όλες τις πτυχές της πολιτικής που απασχολεί την Επιτροπή μας, αλλά και πρακτικές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η Επιτροπή σε καθημερινή βάση. Η γραμματεία, ο ρόλος των πολιτικών ομάδων, των συμβούλων και πολλά άλλα. Εάν λοιπόν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες και για την πολιτική και για την Επιτροπή μας, η γραμματεία είναι στην διάθεσή σας ανά τελειώσαμε και με την τρίτη ανακοίνωσή μου. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, εάν δεν υπάρχουν σχόλια. Σημείο 4 είναι η επιβεβαίωση του χρόνου χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων για το 2009. Και αυτό το έχετε στους φακέλους σας, έχει μοιραστεί. Να ξέρετε ότι εγκρίθηκε ομόφωνα το χρονοδιάγραμμα αυτό από την προηγούμενη βέβαια Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αν ε, δεν έχετε να ζητήσετε καμιά αλλαγή, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Οπότε για το υπόλοιπο του 2009 επικυρώνονται οι ημερομηνίε που έχουμε μπροστά μας. Έτσι δεν βλέπω κανένα να ζητάει καμιά αλλαγή. Οπότε συμφωνούμε. Και τώρα περνάμε στο σημείο 5 που είναι ο προπολογισμό του 2010, τμήμα 3. Είναι βέβαια μια πολύ σημαντική στιγμή μέσα στη χρονιά και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη δουλειά της Επιτροπής μας, το θέμα αυτό. Γι' αυτό και στο μεταξύ η Γραμματεία ετοίμασε ένα σχέδιο για την Πρόεδρο που έχει μοιραστεί και σε εσά. Και εδώ θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δηλαδή έχουμε μια προθεσμία για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης και τις τροπολογίες που θα έχουν κατατεθεί στο μεταξύ στην αρχή της επόμενης συνεδρίασής μας που είναι στις 2 Σεπτεμβρίου. Οπότε ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση γιατί κατάλαβα λίγο και από την Κωνσταντσα Κρέλ και από τον Λάμπερ Ρόι ότι υπάρχουν σχόλια. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Το σημείο 5 δηλαδή, προπολογισμό 2010 τμήμα 3 Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω φυσικά ούτε να καθυστερήσω ούτε να δυσκολέψω εδώ την ε, κατάσταση, αλλά στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή, το σημείο 5, το προπολογισμό και είναι ο προπολογισμό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η δικιά μας αντίδραση αρχικά απέναντι στο Σεβούλιο ήταν αρνητική. Θέλαμε να αλλάξουν τα πράγματα, θέλουμε ο προπολογισμό να επανέλθει στα αρχικά προτινόμενα επίπεδα και να αναγνωριστεί το έργο της Επιτροπής μας. Τώρα η δικιά μου παρατήρηση ευθύ εξ αρχής στο σημείο 4 που είναι το σημείο αυτό παιδί της δικιάς μας της Επιτροπής. Στις αρχές της χρονιάς θέλαμε να ξεκινήσουμε ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα και το διαλέξαμε για τη συνοχή και εξετάσαμε πώς μέσα στα επόμενα χρόνια θα πετύχουμε τη συνοχή όσον αφορά την ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασχοληθούμε και με άλλα σημεία του κόσμου. Βασιστήκαμε δηλαδή, συζητήσαμε για ένα πλαίσιο τριών πιλωτικών προγραμμάτων. Πώς θα έχουμε θετικά αποτελέσματα με τον προπολογισμό που έχουμε στη διάθεσή μας. Το ένα είναι το έρασμος που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση. Δηλαδή και σε περιφερειακό επίπεδο πώς θα στηρίξουμε τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την κατάρτιση Για παράδειγμα, τι γίνεται με τους Ρώμα σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Όμως, δεν υπήρχε γραμμή για το 2010. Αυτό εμεί που θέλουμε είναι και να υπογραμμιστεί περισσότερο το σημείο 4, αλλά και η Επιτροπή, όσο γίνεται πιο γρήγορα, το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, να μας ενημερώσει για το πώς πάει το πρόγραμμα αυτό. Ξεκινήσαμε να το υποστηρίζουμε με τέτοια με τέτοιο ενθουσιασμό και η Επιτροπή είχαμε την εντύπωση ότι το ήθελε. Λοιπόν, θέλουμε και το 2010 να υπάρξει προπολογισμό στα 2 εκατομμύρια ένα πρόγραμμα όπω ε, θέλαμε, αλλά και πληροφορίε πιο συγκεκριμένα για το τι γίνεται με τον ηγετικό ρόλο τη Επιτροπή μα στο θέμα αυτό. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε τα πιλωτικά έργα που είχαμε βάλει στον περσινό προπολογισμό να υποστηριχθούν με κονδύλια. Θα έπρεπε η Κομισιόν να γράψει μια έκθεση να μας πει τι έχει συμβεί ακριβώς και νομίζω πως ε, φέτος επειδή κανονικά τα πιλωτικά έργα είναι διετή δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε νέα έργα, αλλά να δούμε αυτά που ξεκινήσαμε πέρσι και πώς έχει πάει η εφαρμογή τους και μετά να αναπτύξουμε την περαιτέρω στρατηγική μας αφού δούμε τα αποτελέσματα αυτών των πρώτων πιλωτικών έργων. Και νομίζω πως ε, υπ' αυτή την ε, έννοια θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και την ε, γνωμοδότησή μας εδώ πέρα για τον προπολογισμό. Να σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Με ακούτε? Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ε, από όσο ξέρω, εδώ στον ε, προϋπολογισμό του 2010 υπάρχουν δύο πράγματα. Τα έργα του Τζάσπερς και του Εράσμους. Θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Από όσο ξέρω τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέχρι το τελευταίο έτος και μετά η Κομισιόν πρέπει να αναλύσει πώς τα κράτη-μέλη έκαναν τις ε, πληρωμές και ποια θα είναι η επιστροφή των κονδυλίων. Εδώ πέρα όμως μιλάμε όσον αφορά τα Ταμείο Συνοχής ε, για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν έχει κλείσει. Υπάρχουν ακόμα χρονικά περιθώρια για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τα κράτη-μέλη και δεν ε, αναφέρεται εδώ πέρα κουβέντα για την ολοκλήρωση του, του προγράμματος ε, των περιφερειακών ταμείων για τα κράτη-μέλη. Αυτό επηρεάζει τον προπολογισμό του 2010 ή όχι. Ε, δεν αντιλαμβάνομαι την κατάσταση. Βεβαίω, η ερώτησή μου αφορά το 2010, όχι τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών ταμείων 2004-2006 όταν μόλις πέρσι έδωσαν τα κράτη-μέλη τα σχετικά δικαιολογητικά και ακόμα συζητείται αυτό στη σχετική επιτροπή. Ναι, παρακαλώ κάποιος εδώ μπροστά ήταν νομίζω. Ναι, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και το δικό μου ερώτημα συνδέεται άμεσα. Έχουμε εδώ πέρα πληροφορίες συνεχώς για το ότι καθυστερούν τα κονδύλια. Το θέμα είναι ότι τα κονδύλια δεν ε, χρησιμοποιούν ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μας δοθούν κάποιες ε, πληροφορίες. Γνωρίζουμε ποια είναι τα υπόλοιπα στον προπολογισμό και εάν γίνεται η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με την εκτέλεση του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω ουγγρικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ επιτρέψτε μου να πω κάτι για τη διαδικασία συνδιαλλαγής σχετικά με τον προπολογισμό. Τα θέματα που ετέθησαν εδώ από τα μέλη της Επιτροπής ήταν θέματα που ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και στη συνδιαλλαγή. Και από πλευράς Κοινοβουλίου προέβημεν σε μονομερή δήλωση. Σε αυτή τη δήλωση καλωσορίζαμε τα βήματα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία εξασφάλιζαν την επιτάχυση των πληρωμών, ή θα γινόταν προσπάθεια επιτάχυση τουλάχιστον των πληρωμών. Ελήφθησαν κάποιε αποφάσει στην άνοιξη από το Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα. Προτείναμε να ληφθούν και άλλα μέτρα, να γίνουν και άλλα βήματα. Απ' την άλλη χαίρομαι που αυτό το θέμα αναφέρθηκε Δηλαδή ότι δεν αρκεί να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη δαπανούν αυτά τα χρήματα, αλλά θα πρέπει να εστιαστούμε και στην αποτελεσματική χρήση των χρημάτων. Χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα για την επίτευξη των στόχων. Γι' αυτό ανακατανύμαμε αυτά τα χρήματα των φορολογουμένων. Και σε αυτή τη δήλωση επιστήσαν την προσοχή και σε κάτι άλλο. Ότι αυτός ο προπολογισμό τον οποίο επεξεργαζόμαστε πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο κρίσης. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συλλέξει διάφορα σχέδια ενισχύσεως και να βρει σχετικά πόρους. Τεράστια ποσά όμως είναι διαθέσιμα στην πολιτική συνοχής, τα οποία διατίθενται για στόχους που μπορούν να βοηθήσουν να αναδιαμορφωθεί η οικονομία, να μετασχηματιστεί. Το ερώτημα είναι, όλα τα προγράμματα των 100 μελών ταιριάζουν για αυτό το σκοπό. Η κλίμακα, το εύρος των προγραμμάτων που εφαρμόζεται στο επίπεδο 100 μελών είναι πολύ μεγάλο. Τα κράτη-μέλη μπορούν, θα πρέπει να μπορούν να επανεξετάσουν τα προγραμμάτα και να είναι σίγουρα ότι είναι πιο εστιασμένε οι δαπάνε για την αύξηση του ΑΕΠ, για το να στηριχθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, να προστατευτούν θέσει απασχόληση, να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Αυτή η μονομερής δήλωση έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια τη διαδικασίας ε, συνδιαλλαγής. Πληροφορηθήκαμε ότι το Συμβούλιο εξετάζει το ζήτημα, το βλέπει με συμπάθεια, τη δική μας θέση, βλέπει με συμπάθεια τη θέση μας και εφόσον είναι σημαντικότατο θέμα, το Συμβούλιο θα ήθελε να επανέλθει επί του ζητήματος το Σεπτέμβριο. Ενδεχομένως θα υπάρξει και διπλή υποστήριξη για αυτή την προσέγγιση. Από ό,τι γνωρίζω, η φιλοσοφία της Επιτροπής αυτής ταιριάζει με αυτά που σας ανέφερα. Ως εισηγητής θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης. Και νομίζω ότι έχουμε πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το περιθώριο. Υποστηρίζω πλήρως αυτό το κείμενο αυτής τη νομοδοτήσεως, στο σχέδιο κειμένου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, η Επιτροπή Προϋπολογισμού λαμβάνει τους αριθμούς και τις ε, πληροφορίες για το τι ακριβώς γίνεται στα επιχειρησιακά προγράμματα και από εκεί μπορούμε να λάβουμε εμείς τις πληροφορίες. Θα ήθελα όμως να κάνω μια παρατήρηση. Όταν λαμβάνουμε αριθμούς, ε, λαμβάνουμε για τον προϋπολογισμό του 2008 και το 2008 είναι ε, το έτος στο οποίο είχαμε την πρώτη έγκριση πολλών επιχειρησιακών προγραμμάτων και πιθανώς, ε, δεν το γνωρίζετε εσείς όλοι, αλλά θα το γνωρίζετε στις τέσσερις εβδομάδες, ε, πως ε, δεν είναι τόσο απλή η διεκπαιρέωση των προγραμμάτων στις περιφέρειες, οπότε θα ήθελα να σας παρακαλώ να σκεφτείτε πως ο βαθμός απορρόφησης το 2008 δεν ήταν τόσο υψηλός όσο τα επιστημούσαμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια στον προπολογισμό του 2010. Σας υπενθυμίζω πως έχουμε έναν κανόνα των νη συν 2 ή νη συν 3, δηλαδή οι περιφέρειες θα πρέπει να δεσμεύσουν τα κονδύλια ε, των σχετικών προγραμμάτων μετά από δύο ή το αργότερο τρία χρόνια για να μπορέσουν πραγματικά να τα υλοποιήσουν. Ε, οπότε θα πρέπει να διαθέσουν και αυτές τα κονδύλια από τη μεριά τους. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αναβάλουμε συνεχώς ε, προς τα πίσω. Δηλαδή το 2009 τα, τα κονδύλια που δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν δεν μπορούν να εξοδευτούν το 2013. Δεν είναι αυτή κατάσταση και τάξη προπολογισμού. Γι' αυτό θα πρέπει να πιέσουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα να κινηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει εμείς ως Κοινοβούλιο, αλλά απ' την άλλη να διατεθούν και τα κονδύλια αυτά για να μπορέσουν να ξοδευτούν στο κατάλληλο χρονικό πλαίσιο. Και η εμπειρία μου εμένα είναι πως η Κομισιόν ε, έχει μία καλή εικόνα, διαθέτει αυτά τα κονδύλια ε, εγκαίρως και ακόμα και αν δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια την κατάλληλη στιγμή μπορεί να διορθώσει αργότερα με μια συμπληρωματική πληρωμή. Αλλά για να επανέλθουμε εδώ πέρα στην ε, πρόταση αυτή που έχουμε μπροστά μας το Συμβούλιο μέχρι τώρα δεν αντιδρούσε σύμφωνα με αυτά τα οποία ήθελε το Κοινοβούλιο και οι περιφέρειες. Ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια όσον αφορά το ευρωπολογισμό. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε να προβεί σε κάποιο σχόλιο. Ιδεμή, μπορούμε να σα αποστείλουμε όλε τι πληροφορίε ταχύτερο δυνατόν. Θα επιμεληθεί η γραμματεία. Ορίστε, κυρία Σέτερ, έχει το λόγο σύντομα να παρατηρήσω πως οπωσδήποτε θα καταθέσουμε τροπολογίες ως πράσινοι. Θεωρούμε πως ε, πολλά κονδύλια εδώ πέρα δεν ε, ξοδεύονται όσον σε σχέση με σύμφωνα με τους στόχους, με της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής μας, ε, μερικά παραβιάζουν και το δίκαιο περί να μην μιλήσουμε για προστασία του κλίματος κτλ. Οπότε δεν θα προτείνουμε νέες γραμμές του προϋπολογισμού, σε αυτό συμφωνούμε, αλλά αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί ότι τα πιλωτικά προγράμματα είναι πράγματι διαιτητή, πράγματι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να συνεχιστούν δηλαδή. Εμείς είμαστε η ομάδα η οποία το είχε υποστηρίξει αυτό στο παρελθόν, το να συνεχίζονται δηλαδή τα πιλωτικά προγράμματα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, λέει η Πρόεδρος. Άλλα σχόλια. Συμφωνούμε λοιπόν πως η γραμματεία θα φροντίσει να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες και θα σας τις στείλει το των δυνατόν. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω πως ε, όταν η Κομισιόν προετοιμάζει τις προτάσεις ε, προσωρινών δεσμεύσεων και πληρωμών για τα επόμενα έτη χρησιμοποιεί και λαμβάνει υπόψη δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα την ε, τρέχουσα κατάσταση προόδου του κάθε επιχειρησιακού προγράμματος αλλά κοιτάει και την πείρα του παρελθόντος για να μπορέσει να κρίνει. Οπότε συμφωνούμε νομίζω η γραμματεία θα το φροντίσει. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 10 Αυγούστου. Σας το υπενθυμίζω. Ωραία, σας ευχαριστώ. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι τα διάφορα, από ό,τι κατάλαβα. Θέλει κανείς ε, κάτι να πει στα διάφορα? Εάν όχι, λύεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα να ζητήσω από το Προεδρείο και τους συντονιστές να παραμείνουν για την συνεδρία των συντονιστών, για τους υπόλοιπους